Mes chers collègues, à Καθίστε, συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε την συνεδρίασή μας. Επιτροπή των Προϋπολογισμών. La séance est ouverte. Άρχεται η συνεδρίαση. Εάν δεν υπάρχει ένσταση, συνάδελφε, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Επίσης, να σας πω το εξής. Είχαμε κάποιες ε, αλλαγές ε, όσον αφορά τους συντονιστές μας. Ο Τζόρντι Σολέ θα αντικαταστήσει τον Ίντρε Ταρά για το κόμμα των Πρασίνων και ε, ο κύριος ε, Αρνότ αντί του κυρίου Φίντς για το EFDD. Έχετε λάβει τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, Θεωρώ ότι εγκρίνονται. Les points à l'ordre Τώρα, το πρώτο θέμα τη ημερησία διατάξεω αφορά την εκτέλεση του προβολισμού τη κρίση του 2018. Και ακριβώ όπω γίνεται σε τακτά διαστήματα, σε συνεργασία με ε, τον ε, κύριο Μωρεσάν, τον Γενικό Εισηγητή, έχουμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα ο κύριο Ζωάν Ουρέλ, ο οποίο είναι διευθυντή τη Ορμόδας Γενική Διεύθυνση, ούτω ώστε να μπορεί να μα παρουσιάσει μια επισκόπηση του τι γίνεται με την εκτέλεση του προπολογισμού. Αυτό θα γίνει, αυτό αφορά μάλλον το τέλο τη χρήση του 2018 και θα υπάρξει ευκαιρία να μιλήσουμε ακριβώ για ε, το πώ πάνε τα θέματα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμών, αυτονόμων μεταφορών, αποδεσμεύσεων, όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση θα μιλήσουμε για ε, τις πιστώσεις αποδεσμεύσεων, ένα θέμα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα με τις ε, διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό. Και στα πλαίσια αυτά συζητήθηκε ε, κατά πόσο μπορεί να εκτελεστεί να, συγγνώμη, να, να, επικαλεστούμε, να χρησιμοποιήσουμε το 15.3 του καινούργιου δημοσιονομικού κανονισμού. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ουρέλη, τον ευχαριστώ που ήρθε και να δούμε ποιες είναι οι δημοσιονομικές συνέπειες αν δεν υπάρξει ε, συμφωνία για το Brexit. Έχει το λόγο κύριε Ουρέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 18ου. η εκτέλεση πήγε πάρα πολύ καλά, όλα εύρεθμα, ομαλά, για όλα τα προγράμματα, για όλα τα κεφάλαια, τα τμήματα του προπολογισμού. Επιταχύνθηκε η εκτέλεση, οπότε μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει τη χρήση με σχεδόν πλήρη εκτέλεση. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αντίθετα με το 16 και το 17, το 2018 όλα αυτά τα κάναμε χωρίς να χρειαστεί να έχουμε τροποποίηση του προπολογισμού για να μειώσουμε τις ε, πιστώσεις ε, πληρωμών. Θα έχουμε την πλήρη εικόνα όταν κλείσουμε του λογαριασμού στον ε, Μάρτιο. Δεν έχουμε δηλαδή τη σχετική έκθεση, αλλά 99,9% λένε πω οι εκθέσει των υποχρεώσεων εκτελέστηκαν και 99,8% των πιστώσεων ε, πληρωμών. Επομένως αυτό σημαίνει ουσιαστικά πλήρη εκτέλεση. Επίσης, η αναμενόμενη υποεκτέλεση όσον αφορά τις πληρωμές είναι λίγο πάνω από τα 200 εκατομμύρια για όλα τα κεφάλαια του προϋπολογισμού και πάνω από 100 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω, για τα ειδικά εργαλεία. Οπότε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υποεκτέλεση για τις πληρώσεις. Έχουμε κάπου 300 και λιγότερο από πέρσι. Βέβαια, αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία θα τα έχουμε στο σχέδιο του τροποποιητικού προπολογισμού μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία διαμορφώνουν το πλεόνασμα ε, και αυτός ο τροποποιητικός προϋπολογισμός στο σχέδιό του μέχρι 15 Μαΐου θα σας έχει υποβληθεί. Να δούμε τώρα κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής που γνωρίζω ότι ε, ενδιαφέρει πολλούς από εσάς. Όσον αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων 7 ε, έως 17 η πλειονότης ε, των προγραμμάτων αυτής της γενναίας τώρα ε, έχει ολοκληρωθεί, είναι ολοκληρωμένα τα προγράμματα. Αρχάς του 2018 είχαμε σχεδόν 12 δις από εκκρεμούσες ε, υποχρεώσεις, τα RAL δηλαδή, αρέστα λικιντέ και άρα τέλος του 18 είχαμε συρρήγνωση 4,8 δις για την προηγούμενη γενιά των προγραμμάτων. Τώρα, για τη φετινή χρονιά περιμένουμε οι τελευταίες σημαντικές πληρωμές για τα προγράμματα 7 έως 13 πρόκειται να γίνουν το 19 και ό,τι απομείνει στο τέλος του 19 σε μεγάλο ποσοστό θα αποδεσμευτεί. Για να δούμε τώρα τα προγράμματα για την περίοδο 14 έως 20. Όπως γνωρίζετε και θα θυμάστε, η εκτέλεση άρχισε με αργό ρυθμό 14, 15 και 16. Στη συνέχεια από το 17 είχαμε επιτάχυνση και το 18 το σύνολο του εγκριθέντος προϋπολογισμού για το Διορθωτικό Ταμείο και το Ταμείο Επενδύσεων ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ μικρές εξαιρέσει όπως τα 18 εκατομμύρια των πιστώσεων πληρωμών για τους πλέον ε, στερημένους ε, και 99,6% των πιστώσεων πληρωμών έχουν ε, γίνει όσον αφορά διαρθρωτικό ταμείο και ταμείο επενδύσεων. Επίσης θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο σημαντικό, ότι οι δηλώσεις για τις πληρωμές των κρατών μελών ήταν τόσο εκτεταμένες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έδωσε 8 ε, δις από, τα, από τις πράξεις που είχαν προκύψει από την ετήσια εξέταση και καθάριση των λογαριασμών. Επόμενα έχουμε 6,7 δις τα οποία εκταμιεύτηκαν για αυτές τις εισπράξεις, δηλαδή 85% και παραπάνω από το σύνολο, οπότε έχουμε 1,3 δις το οποίο έμεινε αχρησιμοποιητό και μεταφέρθηκε και μπορεί να αξιοποιηθεί στο ενεστός έτος. Φέτος η αξίωση των κρατών μελών σαν αφορά τις πληρωμές προχώρησε αργά μέχρι τον Νοέμβριο. Όμως στη συνέχεια τον Δεκέμβριο είχαμε 18 δις από εφαρμογές πληρώσεων από τα από το 3% ε, των πληρωμών συνέβησαν τον Δεκέμβριο και ήταν σημαντική η προσπάθειά μας, ούτως ώστε όλα αυτά να καλυφθούν και έτσι αυτές οι αξιώσεις ικανοποιήθηκαν πριν το τέλος του έτους και ως αποτέλεσμα ε, έχουμε κρεμούντα συνήθι ποσά 3,4 δις κάποιων εφαρμογών πληρωμών που ήρθαν μετά τις 27 Δεκεμβρίου και άρα δεν μπορέσαμε να τα διεκπαιριώσουμε πριν το τέλος του έτους. Εν τω μεταξύ πάντως τώρα που μιλάμε έχουν αυτές οι αξιώσεις ικανοποιηθεί. Επίσης μετά τις αξιώσεις μετά τις 27-12 έχουμε 1,5 δις πληρωμών, ε, φορολογών πληρωμών που έχουν μπει στην, στην ε, άκρη για να αναλυθούν τέλος πάντων προς το παρόν έχουν ανασταλεί. Σας υπενθυμίζω ε, ο Δεκέμβριος του 2014 ήταν πολύ σημαντική ε, υποθεσμοί γιατί έχουμε τον ΙΣΥΝ 3 για τις αποδεσμεύσεις και στα πλαίσια του αναπρογραμματισμού σε για εκείνη την ε, περίοδο ε, έγινε αναπρογραμματισμός και το 14 πήγε στο 15 επομένως είπαμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αυτό με αποδεσμεύσεις σύμφωνα με τον ΙΣΥΝ οπότε τέλος του 2018 αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν δύο ετήσιες δόσεις αλλά λόγω του ότι είχαμε όλες αυτές τις αξιώσεις το Δεκέμβριο σημαίνει ότι ο στόχος για τις αυτόμες αποδεσμεύσεις επετέχθη. Άρα το μάξιμου ποσό, ούτω ώστε να έχουμε αυτόμετες αποδεσμεύσεις για το τέλος του 2018, πάει μόνο στα 250 εκατομμύρια, το οποίο νομίζω ότι είναι μια καλή επίδοση. Επίσης θα πρέπει να σας αναφέρω ότι η ακρίβεια των προγνώσεων των κρατών μελών έχει βελτιωθεί. Πριν από δύο χρόνια αυτή η ακρίβεια ήταν πολύ μέτρια και ε, το ποσοστό σφάλματος ήταν 48% για όλα τα κρατημέλη. Το 18% η ακρίβεια για το 1β πήγε στο 6%. Άρα πρώτη για τεράστια βελτίωση. Οπότε αυτή η ευξημένη ακρίβεια μας επιτρέπει να βελτιώσουμε ποιότητα και ακρίβεια των δικών μας προγνωστικών των πληρωμών και εκταμιεύσεων. Ε, Επίση έχουμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον καθορισμό των εθνικών αρχών. Τέλος του 2018 απέμειναν μόνο δύο λειτουργικά προγράμματα για τις καθορισμένες ε, αρχέ που έπρεπε να υπάρξει κοινοποίηση. Άρα έχουμε σύνολο 564 και αυτό αφορά ένα πρόγραμμα για τους πιο αποστερημένους το Ηνωμένο Βασίλειο και το λειτουργικό πρόγραμμα για το Σεν Μαρτέν στη Γαλλία το οποίο λόγω της ε, Ήρμα, του, του, του τυφώνα, του κυκλώνα ε, πήγε πίσω. Άρα ε, γι' αυτό κολλήσαν τα πράγματα όσον αφορά την εκτέλεση παλιά τα πρώτα χρόνια. Ε, τώρα ολοκληρώθηκε το ζήτημα. Και τώρα τα, το ΕΣΥΦ, η συνοχή τέλο πάντων, είναι στο 27% της εκτέλεσης για αυτή την ε, επταετία σε σχέση με το 16% τέλους του περασμένου έτους και 9% τέλους του 16%. Όσον αφορά τη συνοχή, ολοκληρώνουμε λέγοντας ότι άλλο ενθαρρυντικό είναι ότι το ποσοστό της επιλογής έργων στα κράτη-μέλη επίσης ε, προόδου πήγε μπροστά το 18 ε, πήγε καλύτερα και πάμε τώρα στο 67% σε σχέση με το 44% πριν από ένα χρόνο. Και αφού έχουμε 27% εκτέλεση και 67% είπαμε για την επιλογή, αυτό σημαίνει ότι πολλά έργα βρίσκονται καθοδόν και αυτό σημαίνει ότι στο προβλεπόμενο μέλλον θα έχουμε καλή εκτέλεση. Να σου πω τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τι αυτόνομε αποδεσμεύσει, αυτόνομε μεταφορέ πιστώσεων. Εμεί χρησιμοποιούμε αυτέ τι αυτόνομε μεταφορέ πιστώσεων. Ε, τι χρησιμοποιούμε αρκετά στα πλαίσια βέβαια του κανονισμού, τόσο ώστε να έχουμε πιο ομαλή εκτέλεση του προπολογισμού. Οι περισσότερε από αυτέ τι ε, μεταφορέ αφορούν προσαρμογή στι λεπτομέρειε των αναγκών χρηματοδότηση. Πολύ πολύ λιγότερο οι αυτόνομε μεταφορέ χρησιμοποιούνται για τις υποχρεώσεις και να σας πω κάποια παραδείγματα χτυπητά για πέρσι. Στο 1β, στο 1β είχαμε κάποιες υποχρεώσεις που έπρεπε να, ε, να αλλάξουν ε, περιφέρεια ή κατηγορία και μεταξύ Κοινωνικού Ταμείου και Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ούτως ώστε να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τις υποχρεώσεις με τις μεταβολές όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα λειτουργικά προγράμματα των κρατών μελών. Άλλο παράδειγμα είναι το κεφάλαιο 4 του προπολογισμού. Μετακινήσαμε 23 ε, εκατομμύρια από το IPA στο ΙΕΝΕ για σε σχέση με το Μαρόκο. Και αυτό κατέστη εφικτό διότι είδαμε ότι έχουμε ε, εισπράξεις ε, κατεχωρημένες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Οπότε θα έπρεπε να δούμε για το IPA αν θα υπάρξουν συνέπειε. Επίσης για το τμήμα κεφάλαιο 3, εκεί που είχαμε την υπηρεσία συνοριοφυλακή και εκτοφυλακής και εκεί έγινε περικοπή στον υπολογισμό, οπότε μπορέσαμε να μεταφέρουμε στην Άμυφ, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε για την κατεπίγουσα βοήθεια περισσότερη πρικοδότηση. Επίση, υπενθυμίζω, είχαμε αυτόνομη μεταφορά για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προβλέπει ο Δημοσιονομικό Οργανισμό για μα. Ε, όποτε υπάρχει κάποια κρίση μετά την πρώτη Δωδεκάτου. Στις 20 Δωδεκάτου πέρσι η Επιτροπή σε αυτά τα πλαίσια ανέπτυξε και πάλι και εκταμείευσε 10 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια υποχρεώσεις και πληρώμες αντίστοιχα για κάποιες υποχρεώσεις που δεν χρησιμοποιηθεί για το 4 όσον αφορά την ανθρωπιστική αρρωγή για να μπορέσει να αυξήσει την βοήθεια, την προκοδότησή της τέλο πάντων για την συνεχιζόμενη κρίση στην Ιεμένη όπως τα προβλέπει ο κανονισμός η αρχή του προπολογισμού Βεβαίως ενημερώθηκε εσείς. Ε, σήμερα σε λίγη ώρα πρόκειται να κάνετε τη σχετική ψηφοφορία ε, για αυτές τις μεταφορές πιστώσεων. Αυτό ήταν περιορισμένο φέτος και έχουμε την μεταφορά 64 εκατομμυρίων από το κεφάλαιο 4 προς την ενίσχυση ε, των κάποιων αναπτυξιακών προγραμμάτων για να καλύψουμε ό,τι χρειάζεται και να επιστρέψουμε κάποια χρήματα ε, στα κράτη-μέλη για κάποιο συνδιαχείριση που, όπου ε, κρεμούσαν αυτές οι πληρωμές. Τώρα όσον αφορά το, τις αποδεσμεύσεις το σύνολο, το σύνολο τους για το 18 φτάνει στο 2,5, 2,5 δις. Αυτό είναι χαμηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Πέρσι είχαμε 5,3, πριν από δύο χρόνια 3,7 δις. Και συγκεκριμένα το ποσό που αποδεσμεύτηκε για το 1β είναι πολύ λιγότερο από όσο πέρσι. Το 17 αποδεσμεύσαμε γύρω στα 3 δις για το 1β. Κυρίως για να κλείσουμε τα προγράμματα 7-13 την προηγούμενη γενιά φέτος οι αποδεσμεύσεις για το 1β είναι λιγότερο από 0,4 δις και για τα άλλα κεφάλαια του προπολογισμού έχουμε κάποιες διαφοροποίησεις ε, αιτήσει αλλά οι υποδεσμεύσει του 18 ευθυγραμμίζονται με την τάση των προηγουμένων χρήσεων. Όσον αφορά τώρα την αποδέσμευση ή τις αποδεσμεύσεις, το τι διατίθεται δυνάμει του 15.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Το 18 είχαμε 281 εκατομμύρια ε, αποδεσμεύσεων για την έρευνα έγιναν αυτό έγινε δυνάμει του 15. Άρα έχουμε λίγο μικρότερο ε, ποσό, γιατί είχαμε 4 εκατομμύρια και κάτι ε, πέρσι, που το συζητήσαμε σε τόσο ζωηρή συζήτηση ε, πέρσι. Και επίση με τις εκθέσεις μας καλύπτουμε τώρα και αυτό το ποσό πια. έχω ολοκληρώσει. βεβαίω και πρόκειται να έχουμε κάποια έκθεση που κατά θα τα λέει και επίσης μια αξιολόγηση ενδελεχής θα σας παρουσιαστεί στα πλαίσια της έκθεσης προβλέψεων, της έκθεσης Άβλη. Αυτά θα ζητηθούν όσον αφορά τις συνεδρίες που θα κάνουμε για τι πληρωμές που προβλέπεται να γίνει στι 20 Μαρτίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για τις διευκρινήσεις. Ο Γενικός Συγητής κ. Μορεσάν επιθυμεί να κάνει παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Διευθυντή για τις παρατηρήσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους για την πολλή δουλειά που έκαναν μαζί μου για να καθορίσουμε προτεραιότητες του προπολογισμού, έγκρισή του στο Κοινοβούλιο, να προχωρήσουμε με επιτυχία στον τριμήρη διάλογο με τα δύο άλλα θεσμικά όργανα και να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προπολογισμού. Θεωρώ ότι ο προπολογισμό του 2018 σε ό,τι αφορά την εκτέλεσή του ήταν ο καλύτερος προϋπολογισμός από τότε που άρχισε το 2014 το παρόν ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε βάλει δηλαδή σωστέ προτεραιότητε, έχουμε εντοπίσει μαζί με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα που πρέπει να διατεθούν τα χρήματα και τα χρήματα επίσης τα κονδύλια δηλαδή απορροφήθηκαν, όπως εξήγησε ο Διευθυντής, με σωστό τρόπο. Πρόκειται για το πέμπτο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και έτσι μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον. Ήταν καλό που ήταν εξαιρετική, εξαιρετικά καλή η εκτέλεση του προπολογισμού. Σωστό θα είναι να είναι το ίδιο καλές οι εκτελέσεις και των επόμενων προϋπολογισμών από 1η Ιανουαρίου 2021, με το νέο δηλαδή ΠΔΠ. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ το δυνατόν συντομότερο και στη διαπραγματεύση με το ε, Συμβούλιο και βεβαίω και με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ιδίω ενθαρρυντικό ήταν το επίπεδο των πληρωμών στο 1β που φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους των προγραμμάτων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό κονδύλια που Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπολογισμό αυτό τα πήγε πολύ καλά στην εκτέλεση. Εντοπίστηκαν οι σωστέ προτεραιότητε και σε συνεργασία με τι χώρε μέλη διασφαλίζουμε ότι τα κονδύλια θα φτάσουν στου δικαιούχου. Μια συγκεκριμένη ερώτηση ό,τι αφορά τι αποδεσμεύσει και υποχρεώσει οι οποίε μεταφέρονται από το 2018, στο 2018 από προηγούμενα χρόνια. Εάν συγκρίνουμε τις αποδεσμεύσεις με το επίπεδο των συνολικών δεσμεύσεων, το ποσό είναι σημαντικό. Αναφέρω για το COSME, για παράδειγμα, 55 εκατομμύρια αποδεσμεύσεις. Οι συνολικές υποχρεώσεις για το 2018 ήταν 354 εκατομμύρια. Ποσά δηλαδή υποχρεώσεων τα οποία μεταφέρονται από έτος σε έτος. Για τις μεταφορές, 281 εκατομμύρια αποδεσμεύσεων ενώ ήταν 1,89 δισεκατομμύρια οι συνολικές ε, υποχρεώσεις. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί από τα ποσά των υποχρεώσεων σημαντικό μέρος αποδεσμεύτηκε. Αυτή είναι η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω και την συνδυάζω με την ερώτηση που υπέβαλα. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προπόρισμού και τις και τους συναδέλφους για την συνεργασία τους. Λίγοι εδώ η εργασία μας πλέον για τον προπολογισμό του 2018 και με την μεταφορά που θα εγκρίνουμε σήμερα το πρωί βάζουμε την τελευταία σφραγίδα στον, ε, στον, στον του 2018 και θα προχωρήσουμε πλέον στον ε, ε του 2019. Ευχαριστώ κύριε ε, Γενικέ Ισηγητά. Ο πρόεδρος, έχω μια διευκρίνηση. Αποδεσμεύσεις 2018 για πιστώσει 2018. Δεν υπάρχουν δηλαδή αποδεσμεύσει για υποχρεώσει που είχαν αναλυφθεί από προηγούμενα χρόνια. Α διευκρινίσει ο κύριος Κουρέλ, Ουρέλ. Συγγνώμη. Και επίση με την ευκαιρία μπορείτε να επιβεβαιώσετε την δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ε, εφημερίδα Πολίτικο, διότι στη δήλωση αυτή λέγεται ότι η εφαρμογή του προϋπολογισμού 2019 θα επιβραδυνθεί σχετικά με δηλώσεις για την μοίρα της συμφωνίας ή της έλλειψης συμφωνίας. αλλιώτικο από αυτό που είπε ο κ. Σελμάιερ, που είναι ο Γενικός Γραμματεύς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνάντηση την οποία οργανώσαμε στο Στρασβούργο, που είχε δηλώσει ότι οι Βρετανοί θα ε, σεβαστούν τις νομικές τους δεσμεύσεις. Θα θέλαμε κάποια διευκρίνηση σχετικά. Εσείς κύριε Ουρέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γενικό Εισηγητή για την ερώτησή του. Για την συγκεκριμένη ερώτηση του κύριου Μουρεσάν, νομίζω ότι χρειάζεται λεπτομερής απάντηση γραπτός, την οποία θα συντάξω και θα σας διαβιβάσω σύντομα. Όσον αφορά τις ερωτήσεις του Προέδρου επιβεβαιώνω ότι όχι σε μεγάλο βαθμό οι αποδεσμεύσεις που έγιναν το 2018 απηχούν δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί το 17, 16 και 15. Για παράδειγμα, οι περισσότερες από τις αποδεσμεύσεις συνοχής προέρχονται από προηγούμενα προγράμματα, προηγούμενη γενεά προγραμμάτων. Το λέω αυτό εκτός βέβαια εάν παρενόησα την ερώτησή σα, Όχι, καλά την καταλάβατε, απαντά ο πρόεδρο, για να καταλάβουμε καλά τι εννοούμε. Οι πιστώσει του προπολογισμού 2018 και οι αποδεσμεύσει μπορούν να αναφέρονται στους προπολογισμού 16 έω 18 ή και παλαιότερα, απαντά ο κυριο Σουρέλ. 2007, 2007-2008. Άρα δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στον προπολογισμό 2018 και στις αποδεσμεύσεις. Οι αποδεσμεύσει αναφέρονται σε προηγούμενους προπολογισμού και το ποσοστό που παρατηρούμε θα πρέπει δηλαδή να αναλυθεί για να γνωρίζουμε ακριβώς εάν είναι από προηγούμενα έτη ή όχι. Διότι το αντιλαμβάνομαι ως μια διόρθωση που γίνεται στον προπολογισμό του 18, αλλά φαίνεται πως δεν συμβαίνει αυτό. Είναι αποδεσμεύσεις σε σχέση με υποχρεώσεις που είχαν αναλυθεί επί προηγουμένων προπολογισμών. Σωστό θα είναι στο μέλλον όταν διαβάζετε τη σχετική πληροφορία να το κάνετε γραπτός και να μας λέτε καθαρά οι αποδεσμεύσεις ποιον προϋπολογισμό αφορούν. Απάντηση του Διευθυντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα το σημειώσω αυτό. Είναι σχετικά απλό να σας παράσχουμε μια ανάλυση για τις αποδεσμεύσεις που έχουν γίνει ε, μέσα στο παρόν πι και αποδεσμεύσεις που έχουν γίνει από το προηγούμενο πι γιατί γίνονται από ξεχωριστά, ξεχωριστές γραμμές του προϋπολογισμού. Μπορεί λοιπόν να σας δοθεί αυτό σχετικά εύκολα, αλλά για επιμέρους χρόνια, επιμέρους έτη δηλαδή, ε, είναι πιο δύσκολο. Θα κοιτάξουμε αν είναι εύκολο να γίνει αυτό που ζητάτε. Επανέχει το Πρόεδρος. Ο Γενικό Εισηγητή μα είπε πριν ότι ο προπολογισμό του 2018 ήταν καλά συνταγμένο και οδήγησε σε σχετικά λίγε αποδεσμεύσει. Αν κατανοώ καλά, οι αποδεσμεύσει αυτέ δεν αναφέρονται στο 2018, αλλά σε προηγούμενα έτη. Μουρεσάν. Πρόκειται για αποδεσμεύσει ποσών από προηγούμενα χρόνια, τα οποία μεταφέρθηκαν προ τα εμπρό. Το ποσό είναι σημαντικό σε αναλογία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 2018. Αυτό ρωτώ. Και ε, χαίρομαι που δεσμεύτηκε ο κύριος Διευθυντής ότι θα υποβάλει απάντηση γραπτός. Είναι από προηγούμενους προϋπολογισμούς, δεν αναφέρονται στον 2018. Αλλά είναι σημαντικό για μας ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να το γνωρίζουμε γιατί είναι σημαντικά τα ποσά σε σχέση με τις πιστώσεις ενός έτους και το 2018 το πήρα ως έτος αναφοράς. Σύμφωνοι, λέει ο πρόεδρο. Τώρα για το πολίτικο, για την εφημερίδα πολίτικο, τι έχετε να πείτε. Απάντηση. Ας διευκρινίσουμε μία ενδεχόμενη παρανόηση. Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να λάβει ένα καθαρά εσωτερικό μέτρο προφύλαξης. Δώσαμε στους authorizing officers στην παρούσα περίοδο του προπολογισμού το 85% των πιστώσεων. Αυτό με κανένα τρόπο δεν σημαίνει επιβράδυνση της εφαρμογής του προπολογισμού. Το 85% αρκεί και με το παραπάνω για όλους τους authorizing officer να προχωρήσουν με την ε, φυσιολογική εκτέλεση του προπολογισμού και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπου κατ' εξαίρεση είναι αναγκαίο να διατεθούν το 100% των πιστώσεων, όπως για παράδειγμα στη συνοχή, εδώ ήδη έχει διατεθεί το 100%. Για να είμαι σαφής λοιπόν δεν υπάρχει απολύτως καμία διάθεση, καμία πρόθεση καλύτερα να επιβραδυνθεί η εκτέλεση του προπολογισμού. Πρόκειται για καθαρά προφυλακτικό μέτρο και αυτή τη στιγμή σε αυτό καταστεί δυνατό. Το υπολοιπόμενο 15% θα διατεθεί επίση στου ε, έχοντε την ε, υπογραφή τη εγκρίση, authorizing officers δηλαδή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο έτερος ε, ζητεί το λόγο και επειδή λίγο έχουμε καθυστερήσει, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, ε, προτείνω να αρκεστούμε σε αυτά. Ευχαριστώ τον Γενικό Εισηγητή κύριο Μούρεσαν. Η παρέμβασή σας ήταν και λίγο συναισθηματικά φορτισμένη γιατί πρόκειται για την τελευταία πράξη του, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ και τον κύριο Ουρέλ. Θα προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες ε, ε, στην κατάλληλη σχισμή της ε, συσκευής σας. Ας κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, λοιπόν για τη δοκιμαστική αυτή ψηφοφορία, όπως εξήγησα. Ξέχασα την κάρτα μου, λέει μία βουλευτής, ε, σε άλλη επιτροπή. Θα νομίζω ότι πρέπει να έχετε χωριστές κάρτες για τις διάφορες επιτροπές, λέει χαριτολογών ο πρόεδρος. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Είδα ότι ορισμένοι ψηφίσατε κατά στη δοκιμαστική. Και ορισμένοι είχατε, είχατε διάθεση για αποχή. Τώρα λοιπόν για την έκθεση του κύριου Κέλμελ. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 Κόλμελ υπέρ κατά αποχές επαλήθευση αρχίζει ηλεκτρονική δηλαδή επαλήθευση πέρας εγκρίνεται 19 υπέρ 11 είστε υπέρ κυρία μου μάλιστα ευχαριστώ Άρα 20 υπέρ. Εγκρίνεται. Άρα η παριθμόν 10 τροπολογία εκπίπτει. Η 11 τώρα. Α, επίσης εκπίπτει. Η παριθμόν 2 ψηφίζεται. Ψήφι υπέρ παρακαλώ, τις δύο, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 εκπίπτει διότι ενεκρίθη 12. 13 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται με ψήφους 15 κατά 14 υπέρ. Α, 15-15. Ισοψηφία. Παρ' όλα αυτά απορρίπτεται. Υπαριθμόν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 5 εγκρίνεται χωρίς ψηφοφορία. Υπαριθμόν 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 7 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά αρχίζει πέρας απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παριθμόν 8 πέρας απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με ψήφους 26 υπέρ, 27 με την κυρία Τόμα, 3 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Κέρμελ. Για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού 2018 της Επιτροπής υπό την ευθύνη του εισηγητού Σίγφριτ Μουρεσάν. Έχουν γίνει, ε, συζητήθηκαν αυτά ήδη στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο ε, Ουρέλ. Έχετε κάποια δήλωση κύριε Γενική Εισηγητά. Σωστό είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για την μεταφορά αυτή με περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι διόλου αμφιλεγόμενοι Είναι προφανής. Συνιστώ στους συναδέλφους να υπερψηφίσουν. Πρόκειται για ένα σύνολο 64 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών που θα μεταφερθούν σήμερα, 25 εκατομμύρια από τον τίτλο 4 για την ε, ολοκλήρωση προενταξιακών ε, στηρίξεων για έργα στην Τουρκία. 25 εκατομμύρια ευρώ πάλι από τον τίτλο 4 για την ολοκλήρωση δράσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας λόγω καθυστερήσεων κάποιων ε, πληρωμών στο Μαρόκο. Θα μεταφέρομαι 10 εκατομμύρια ευρώ από τον τίτλο 4 DCI ασφάλεια τροφίμων λόγω της καθυστερημένης ε, έγκρισης του ετησίου σχεδίου 2018 που οδήγησε σε ορισμένες καθυστερήσεις πληρωμών, 3,2 εκατομμύρια από τον τίτλο 4 μελέτες για την δομή γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πάλι διότι το συνολικό επιλέξιμο κόστος ήταν χαμηλότερο από το ανώτατο δυνατό επιλέξιμο κόστος. Και τέλος, 0,8% από τον τίτλο 2, από τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές για το 2019. Άρα συνολικά 64 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μεταφερθούν στο Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου. Για, πρόκειται για δαπάνες του τρίτου τριμήνου του 2018. Αυτή είναι η μεταφορά που συνιστώ και παρακαλώ τις και τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν. Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά. Ποιος επιθυμεί να τοποθετηθεί. Εσείς κύριε Διευθυντά δεν υπάρχουν σχόλια. Άρα, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ας ψηφίσετε λοιπόν, αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι, όχι ακόμη. Θα κλείσουμε όμως τώρα την ψηφοφορία. Έγκριση, 26 ψήφοι, 27 κυρία Τωμά, 27 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές, μάλλον συγγνώμη, δύο ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια κύριε Γενικέ Εισηγητά για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού 2017. Δεν υπάρχουν ε, αιτήματα μεταφοράς. Το λόγο λαμβάνει ο κύριος Πολ Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία επιθυμία μεταφορών από το ελεγκτικό συνεδρίο το οποίο επιθυμεί να ε, ε, ιδρύσει δύο ε, θέσεις μονίμων βοηθών. Το ελεγκτικό συνέδριο θα κάνει την σχετική τροποποίηση του οργανογράμματός του στις επόμενες τρεις εβδομάδες και τάσσομαι υπέρ της σχετικής μεταφοράς. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Άρα, θεωρώ ότι εγκρίνεται η αίτηση μεταφοράς. Τώρα η κυρία Χολμπάιερ, διαρκής εισηγητής για την πολιτική κτίριων. Ε, θα μας εξηγήσει τα σχετικά με ένα κέντρο καλωσορίσματος του Μπερλεμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα οικοδομικό έργο, το οποίο θα είναι το λεγόμενο Welcome Center του κτηρίου Μπερλεμό, όπως και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ωραίο τίτλο σε, στην πραγματικότητα εγκαταστάσεις ασφαλείας. Αυτό που ενδιαφέρει εν προκειμένου είναι οι επισκέπτες να μην υφίσταται τον έλεγχο ασφαλείας εντός του κτηρίου Μπερλεμού αλλά σε παράρτημα που θα κτιστεί εκτός, ώστε να είναι ασφαλές το κτίριο Μπερλεμού. Θα είναι ένα ε, Welcome Center 370 τετραγωνικών μέτρων ε, θα έχει σχετικές εγκαταστάσεις ασφαλείας θα αρκεί για έναν αριθμό 90.000 επισκεπτών το κτίριο Μπερλεμό έχει ιδιαίτερη σύμβαση με το βελγικό δημόσιο ε, υπό τη μορφή εταιρείας τότε δεν επιτρεπόταν να δανειστεί ένα θεσμικό όργανο να κτίσει και μετά να αποπληρώσει. Χρειαζόταν λοιπόν συμβάσεις με την συγκεκριμένη χώρα μέλος, εν προκειμένου το Βέλγιο, για να χρηματοδοτηθεί μετά με τη συνεργασία τραπεζών και από την πλευρά δηλαδή του, του, του κράτους και μετά το θεσμικό όργανο να το ε, μισθώσει, να, κάνει δηλαδή μίσθωση μακρού χρόνου, leasing. Έμαθα τώρα και τι σημαίνει, και τι σημαίνει ε, εμφυτευτική σύμβαση. Ε, για πρώτη φορά το άκουσα. Ε, αντιλαμβάνομαι πάντως ότι είναι λογικό αυτό, δηλαδή στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εμφανίζεται πλέον ως κύριος του ε, ακινήτου με 600 τετραγωνικών μέτρων περίπου, όπου μπορεί επ' αυτού να κατασκευάσει, να οικοδομήσει δηλαδή το κέντρο που επιθυμεί. Η σύμβαση με το βελγικό κράτος παραμένει ως έχει, το μίσθωμα δεν αυξάνεται, εμείς πληρώνουμε την κατασκευή του κτηρίου και από το 2031 θα μεταφερθεί η κυριότητα του κτηρίου έναντι ενός ή δύο ευρώ. Πρόκειται για συμβάσεις οι οποίες είχαν λάβει τη μορφή αυτή τότε προετών λόγω των δημοσιονομικών διατάξεων που δεν επέτρεπαν σε θεσμικά όργανα να ε, δανειστούν από τράπεζες. Το ποσό που προβλέπεται είναι 4,29 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει προκήρυξη διαγωνισμού. Ήδη έχει γίνει ο διαγωνισμός. Έχει κερδίσει ο όμιλος επιχειρήσεων Λουίς Τεουάλε. Θα αρχίσει σύντομα η κατασκευή. Αρχικά είχαμε πει ότι η αύξηση του κόστους είναι φυσιολογική, δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτε περισσότερο. Απαλλάσσεται των φόρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών θα υπάρχουν, ε, υπάρχουν τα, οι δαπάνες 8.000 για το ηλεκτρικό ρεύμα, 15.000 για την καθαριότητα αναμήνα. Και βρίσκω ότι τα κονδύλια αυτά είναι μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού, δεν σημαίνουν κανένα κίνδυνο για τον προϋπολογισμό, για υπερβασή του και συνιστώ έγκριση. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία ονομαστική. Αρχίζει. Πέρας. Έγκριση. Ψήφι 27 υπέρ, μαζί με την κυρία Τωμά δηλαδή, 2 κατά. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Τώρα το βασίλειο του Βελγίου εμένει, διότι κάποτε δεν γνώριζαν πού να εγκαταστήσουν τα κτίρια. Το... Είχαν επιλέξει τότε την τοποθεσία του Μπερλεμό, αλλά φαίνεται πως άρεσε τελικά και παρέμεινε ε, σωστή λοιπόν η ε, ε, πρωτοβουλία εκείνη. Άρα έχουμε ολοκληρώσει τώρα την διαδικασία ψηφοφοριών. Το λόγο κρατεί η κυρία Μόνικα Χολμάιρ για να μας εξηγήσει τα του κτηρίου Ήλιος, Χέλιος, το πρώην κτίριο Ντρόσμπαχ και το κτίριο Λακολίτ στο Λουξεμβούργο. Σύντομη πληροφορία. Η μετακόμιση από το κτίριο της Κομισιόν Ζαμονέ θα καθυστερήσει για τεχνικούς λόγους, ώστε οι συμβάσει μισθώσεως των δύο κτιρίων θα πρέπει να παραταθούν. Γίνονται διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ε, συμβάσεις, ώστε να ε, διατηρηθούν οι συμβάσει μισθώσεως μέχρι την ημερομηνία των ε, μετακομίσεων. Αυτοί που εγκαθίστανται στο κτίριο Χέλιος είναι 886, 886 άτομα και είναι διευθύνσεις όπως μετάφρασης ανθρωπίνων πόρων κλπ. Θα μας υποβληθεί ο σχετικός φάκελος τις επόμενες ημέρες, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου και θα διαβιβαστεί με όλες τις λεπτομέρειες και στους κοιότητες εισηγητές και θα ακολουθήσει και συνάντηση με τους εργαζομένους του Λουξεμβούργου για να ρυθμίσουμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια, λέει ο πρόεδρος. Στρέβομαι στον, στους σκιώδεις εισηγητές, αν επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Υπάρχει σκιώδης εισηγητής ή εισηγήτρια που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Κύριε Συγγήτρια, φαίνεται ότι τους πείσατε με τα λόγια σας. Πέραν τώρα των σχεδόν εισηγητών, άλλος κανείς, σχόλια, παρατηρήσεις. Έχει καλώς. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο τι τυπλοφορείται. Μάλλον προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και ειδική έκθεση για τους γραφειακούς χώρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα παρατείνεται η συζήτηση των δύο εκθέσεων της κυρίας ε, Χόλμαϊερ. Καλωσορίζω τα δύο μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, τα οποία παρέχουν, δηλαδή, οι οποίοι ε, είναι παρόντες. Γιάνν Γκρέγκορ, Επίσης παρόντες είναι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων που αναφέρονται στην ειδική έκθεση. Εκ μέρους του Κοινοβουλίου Γενικοί Διευθυντές Ινλό και Φίνς, κύριοι Ινλούς και Κλετή, της Κομισιόν, Ινλό και Μπεκέτ, του Συμβουλίου, η κυρία Βαν για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο κύριος Σμίρς, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Κισελεύσκη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκρεγόρ. Παρακαλώ 10 15 λεπτά για παρουσίαση της ειδική εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την κτηριακή πολιτική της Ενώσεως. Έχετε το λόγο κύριε Γκρεγόρ. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους αντιπροέδρους και τα μέλη της ε, Επιτροπής σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ειδική αυτή έκθεση του ανεκτικού συνεδρίου του προηγούμενου Δεκεμβρίου. σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα και τα σχετικά γραφεία. Να ξεκινήσω και να δομήσω μάλλον την ε, παρουσίασή μου σε πέντε πυλώνες. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι έχει γίνει στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τα θέματα των γραφείων. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσω το πεδίο εφαρμογή ε, του ελέγχου και τέλος θα εστιαστώ και στις παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε και στις συστάσεις. Στο παρελθόν λοιπόν εστιαστήκαμε στις δαπάνε των θεσμικών οργάνων για τα κτίρια το 2007. Είχαμε μια ειδική έκθεση η έκθεση αυτή περιλαμβάνει συστάσεις ε, για τον καλύτερο ορισμό και συντονισμό του πολιτού πλαισίου για τα κτίρια. Επίσης, ε, προτείναμε και συστήσαμε να μετακινηθούμε προς μακροπρόθεσμες ε, μισθώσεις και ενδεχομένως και σε αγορές των κτιρίων. Επίσης, εκτίμηση των αναγκών και της διαχείρισης πληροφοριών έλεγχος της αγοράς και ανταγωνισμός και επίσης τη χρήση φορολογικών απαλλαγών υπό το πρωτόκολλο για τα προνομία και τις ασυλίες. Και τέλος, διαθεσμική συνεργασία. Σε τρεις τομείς ε, θέλαμε να υπάρξει βελτίωση. Υπήρχε καλό επίπεδο με τη διαθεσμική συνεργασία και ότι υπήρξε πραγματικά μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τη μίσθωση ή αγορά των κτηρίων. Τώρα κινηθήκαμε προ την αγορά. Επίση, το 2014 εστιαστήκαμε στην αποκέντρωση των λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης για την έμπρεση εξωτερικής δράσης και τα γραφεία της σε όλο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δαπάνες σε σχέση με τα κτίρια κατά τον ετήσιο έλεγχό μας. Θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα. Το 2010 και στη σχετική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου επισημάνομαι ότι 235 εκατομμύρια ευρώ ε, πληρώθηκαν, προπληρώθηκαν για τα πρώτα τρία χρόνια του κτηρίου Europa και αυτό ε, σε ό,τι αφορά και την πρόοδο του κτηρίου, την έκθεση του 2017 επισημάναμε κάποιες αδυναμίε σε ό,τι αφορά τη δικασία προκήρυξη διαγωνισμό για δύο συμβάσει εργασία για κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκ δεν έχουμε αναφέρει περαιτέρω τέτοια ζητήματα συμμόρφωση στην εκθεσή μας. Θα ήθελα να σα εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα, να σα εξηγήσω και γιατί κάναμε την ε, έλεγχο αυτό γιατί το, οι στα κτίρια είναι 11% του συνολικού διοικητικού προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου ένα δι Αυτό το ποσό είναι μάλλον σταθερό τα τελευταία πέντε χρόνια. Πριν από το διάστημα αυτό όμω ήταν πιο υψηλό. Άρα, μακροπρόθεσμα υπήρξε μείωση. Περίπου 7% έχει να κάνει με μισθώσεις και αγορέ και 4% σχετίζεται με άλλε κτηριακέ δαπάνε όπω η συντηρήση, η ασφάλεια, ενέργεια κτλ. Και φυσικά λάβαμε υπόψη και την αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού του 2013 όπου υπήρξε αυτή η προδιαγραφή για αιτήσει εκθέσει για τα κτίρια και η ικανότητα, δυνατότητα ε, άμα χρηματοδότησης με άμεσες μισθώσεις. 26% λοιπόν ήταν η αύξηση σε σχέση με το 2004 σε ό,τι αφορά τα τραγωνικά μέτρα. Και είχαμε αύξηση προσωπικού κατά 20%. Να σας εξηγήσω ποιο ήταν το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου. Εστιαστήκαμε στα γραφεία, στις γραφειακές καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου 70% της συνολικής έκτασης των θεσμικών οργάνων των κτηρίων. Και γι' αυτό λοιπόν εστιαστήκαμε σε πέντε κτίρια. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή, τα κτίρια και τα γραφεία. Έχουμε λοιπόν γραφεία στις Βρυξέλλε, Λουξεμβούργο και Φραγκφούρτη. Και εστιαστήκαμε ιδιαίτερα σε αγορές και μισθώσεις. Αυτό είναι στα δύο τρίτα των δαπανών των κτηριακών. Δεν κοιτάξαμε τι δαπάνε σε ό,τι αφορά τη συντήρηση, την ασφάλεια, τον καθαρισμό, την ενέργεια κτλ. Όπου υπήρχε δυνατότητα, προσπαθήσαμε να, να συγκρίνουμε με άλλα θεσμικά όργανα και τι πρακτικέ που ακολουθούνται εκεί σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση, την ΕΤΕΠ, το Ελεκτικό Συνέδριο τη Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. για να προσπαθήσω να σας περιγράψω ποια θέματα εξετάσαμε στον έλεγχο. Τι ρωτηθήκαμε καταρχάς, κατά πόσο οι δαπάνες για τις κτηριακές και τα γραφεία τη σωστής και αποδοτικής διαχείρισης. Και τρία είναι τα υπερωτήματα που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή, κατά πόσο υπάρχουν ε, καθιερωμένες στρατηγικές για τα κτίρια για τη συνεργασία για να πετύχουμε περικοπή του κόστους Επίσης εξετάσαμε το πώς ε, αποκτούν ε, τα θεσμικά όργανα, τα γραφεία τους, κατά πόσο γίνεται αυτό με αποτελεσματικό τρόπο δηλαδή. Και επίσης παρακολουθήσαμε και κάναμε αναφορές σε ό,τι αφορά, αφορά τα χαρτοφυλάκια γραφείου, γραφείων. Συλλέξαμε λοιπόν πολλά αριθμητικά στοιχεία, διάφορα ερωτηματολόγια, εκθέσεις, μελέτες, και συνολικά διαπιστώσαμε ότι τα θεσμικά όργανα διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τι δαπάνε αυτέ, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωση σε κάποιου τομεί. Άρα μπορούν να, να βελτιωθούν κάποιε στρατηγικέ, κάποιο σχεδιασμό. Ε, κάποιε από τι δαπάνε δεν είχαν επίσημη αδειοδότηση των προτέρων και θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχουν συγκρίσιμα σενάρια για τα διάφορα όργανα. Οι αποφάσει τώρα σε ό,τι αφορά τα γραφεία ήταν καλά τεκμηριωμένε, αλλά προφανώ οι διαδικασίε λήψη αποφάσεων είναι περίπλοκε. Έγιναν μεγάλε καθυστερήσει ε, σε ό,τι αφορά την κατασκευή μεγάλων έργων και μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων. Αυτό είχε ω συνέπεια επιπλέον κόστο και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω το θέμα τη παρατηρήση. Να περάσουμε στις παρατηρήσεις. Καταρχάς, ε, όπως είπα και αυτή εξ αρχής, τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται, αλλά μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Με συμμετρικό τρόπο βέβαια χρησιμοποιούνται τα μέσα λήψη αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά τα κτίρια, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης δεν είναι πάντα τυποποιημένε και ενημερωμένε αυτέ οι στρατηγικέ για τα κτίρια. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και σχεδιασμό σενάριων. Και επίσης εντοπίσαμε μια καλή πρακτική στην σκόλπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά ένα rolling over, σε ό,τι αφορά το πολίτης ε, πλαίσιο πολιτικής, σε ό,τι αφορά τον νέου τρόπου συνεργασία. Αυτό συνεπάγεται και φυσικά κόστο για τα θεσμικά όργανα. Κοιτάξαμε κατά πόσον υπήρξαν πλανεκτήματα και πραγματικά ωφέλη από τις ε, νέες πολιτικές. Δεν έχουμε βρει ακόμα τέτοια τεκμήρια για το κατά πόσον υπάρχουν οικονομικά ή άλλα ωφέλη. Και προσωπικά θα ήθελα να πω ότι αυτός ο νέος τρόπος εργασίας ήταν πολύ δημοφιλής πριν από κάποιες δεκαετίες. Τώρα πλέον έχει υποροχηθεί θεωρώ σύστημα. Δεύτερη παρατήρηση. Οι αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, εγκαταστάσεις και τα γραφεία είναι πολύ καλά αλλά η χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη και περίπλοκη. Αναλύσαμε κατά πόσον οι αποφάσεις ε, βασίζονταν σε τεκμηριωμένα στοιχεία, κατά πόσον υπήρχε συνεργασία με τη χώρα υποδοχής και υποστήριξη από τη χώρα υποδοχής. Όλα αυτά ήταν ε, θετικά και προφανώς η υποστήριξη από τα κράτη-μέλη από το, τη χώρα υποδοχής ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα υποδοχή, αλλά και με το καθεκτήριο. Η χρηματοδότηση παραμένει ένα περίπλοκο ζήτημα. Και γι' αυτό λοιπόν ε, επηρεάζει και την διαφάνεια του προπολογισμού. Η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων περιλαμβάνει ε, διαμεσολαβητές και οικονομικούς και κρατικούς δημόσιους, μεταξύ των οποίων και την ΕΤΕΠ. Και οι προκαταβολές δεν ε, αναφέρονται πάντα στου αιτήσει προπολογισμού. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το θέμα τη διαφάνεια του προπολογισμού. Τρίτη παρατήρηση σε ό,τι αφορά μεγάλα έργα, κατασκευέ ε, που επηρεάστηκαν από καθυστερήσει και επιπλέον κόστο. Τέσσερα έργα αναλύσαμε: Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή και Ελεκτικό Συνέδριο. Μόνο ένα από τα μεγάλα αυτά έργα ήταν στην ώρα του και εντός του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά το ελεκτικό συνέδριο. Mm. Α, αλλά τα λακτήρια αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και αυτό προφανώς οδήγησε σε επιπλέον επιβάρυνση και κόστος. Και να εξετάσουμε τώρα τα μεμονωμένα έργα σε ό,τι αφορά το λεκτικό συνέδριο λοιπόν ήταν θετικό το αποτέλεσμα όπου τελικά το έργο έμεινε εντός προϋπολογισμού και εντός προθεσμίας χάρη και στη σειρή συνεργασία με τη χώρα συνεργασία, με τη χώρα υποδοχή, το Λουξεμβούργο. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Και πάλι υπήρχε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, αλλά από την άλλη υπήρχε αρνητική εκτίμηση της συνεργασίας με την χώρα υποδοχής και το Συμβούλιο θα πρέπει να αναγκάστηκε μάλλον να αντιδράσει αυξάνοντας το προσωπικό για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά προφανώς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι καθυστερήσεις προέκυψαν και από απρόβλεπτες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, το εργο κατ' CAD2 του Κοινοβουλίου, πάλι υπήρχε καθυστέρηση με επιπλέον κόστος. Ο βασικός λόγος για την καθυστέρηση ήταν η περιορισμένη εμπειρία του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τέτοια έργα και η αρχική προκήρυξη διαγωνισμού που δεν στέφθηκε με πτυχία και η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να μειώσει την έκταση του έργου, να αλλάξει και τις τεχνικές περιγραφές του κτηρίου και να αυξήσει και το οικονομικά τετράγωνα. Αυτό οδήγησε σε πιο πολύ ανταγωνισμό, προκειμένου να γίνει σεβαστός και ο αρχικός εγχωρισμένος προπολογισμό. Παρ' όλα αυτά ε, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 86 εκατομμύρια ε, επιπλέον κόστος σε μία περίοδο 6 ετών. Αυτό προφανώς ε, είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια το έτος. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το GMO2 συγκεκριμένα, είχαμε καθυστερήσει. Είχαμε 15 χρόνια που χρειάστηκε να φτάσουμε σε συμφωνία ε, με το κράτο του Λουξεμβούργου, γιατί υπήρχαν αμοιβαιότητες σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό των αρχιτεκτονικό, σε ό,τι αφορά τα θέματα της προκήρυξη του διαγωνισμού, σε ό,τι αφορά και τις ε, προπαρασκευαστικές ε, εργασίες στο έδαφος και συνολικά θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπολογίσαμε μάλλον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει επιπλέον κόστο μίσθωση 248 εκατομμύρια λόγω των καθυστερήσεων αυτών και λόγω τη εκένωση του κτηρίου GMO1. Τέταρτη παρατηρήση σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση και την ε, υποβολή εκθέσεων. Δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται. Έχουμε πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά το σκέλος αυτό Ορίζει λοιπόν ο δημοσιονομικός ε, κανονισμός ε, τι πρέπει να γίνει, άλλαξαν οι προδιαγραφές του 2013, αλλά δεν προβλέπεται παρόλα αυτά συγκριτική ανάλυση. Επίσης η ανάλυση μας καταδεικνύει ότι λίγο πολύ οι χώροι γραφείου ανάτομο στα θεσμικά όργανα είναι παρόμοιοι. Αλλά άλλοι δείκτες κόστους ενδιαφέρουν ε, πολύ. Τώρα, να περάσουμε στην τελευταία διαφάνεια. Και να σας πω ποιε είναι οι συστάσεις μας. Προτείνουμε λοιπόν στα θεσμικά όργανα να ενημερώνουν και να τυποποιούν τη στρατηγική συντακτήρια τακτικά και να ε, ενημερώνουν και τα σχετικά έγγραφα εργασία, να, εξα... να αξιολογούν ε, τα έργα για τους νέους τρόπους εργασίας, να αυξήσουν επίσης την διαφάνεια ε, προπολογισμού ό,τι αφορά του μηχανισμού ε, χρηματοδότηση για τα έργα κατασκευή και από το 2017 και μετά είχαμε συστήσει να εξετάσουμε και τις διάφορες ε, εκχωρήσεις για τα κτίρια. Επίσης, συστήνουμε να υπάρχουν σωστές και ε, καλές λειτουργίες διαχείρισης για μεγάλα έργα και μεγάλα έργα ανακαίνησης και τέλος να βελτιωθεί η ποιότητα των ε, ε, δεδομένων και η παρακολούθηση ό,τι αφορά τα θέματα των κτηρίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με τους συναδέλφους μου όλους είμαστε στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκρέγκορ για την ε, περιεκτική σας ε, συνθετική παρουσίαση όσον αφορά την πολιτική για τα ακίνητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Eh bien, je vais maintenant donner la parole. Τώρα, η σκητάλη στον ε, εισηγητή μας. Τον μόνιμο εισηγητή για την πολιτική ανακοινήτων. Όμως, έπρεπε να ε, αποχωρήσει. Άλλος, ίσως ε, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού, και αυτή λείπε. Όποιος στείλει τότε, συνάδελφε ως τις βούλετε. Όχι, κανεί, δεν βλέπω κανείς κάποιος να θέλει ερώτηση. Κύριε Γκρεκορ, κάτι συγκεκριμένο από πλευράς μου. Για αυτό το σκούπισμα, το σιπίν, ραμασάζ. Αντικειμενικά μιλώντας, δεν είναι ό,τι πιο ειλικρινές στα δημοσιονομικά. Γιατί παρουσιάζουμε προϋπολογισμούς με υπερεκτίμηση κάποιων κονδυλίων το οποίο είναι παράπτωμα γιατί δεν αντικατοπτρίζει πιστά την πραγματικότητα και αυτό το κάνουμε συστηματικά. Να, στη σελίδα 25 της εκθέσεώς σας αναφέρεται κάτι σχετικά. για κάποιες ε, προκαταβολές όσον αφορά ε, κάποιες κατασκευές και στα ανάλογα κονδύλια αυτά αντικατοπίζονται στον προϋπολογισμό και γενικά αυτή η πρακτική οδηγεί σε μεταφορά πιστώσεων που φύγει την διαφάνεια και αποτελεί παράβαση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και έτσι ο προϋπολογισμός σε σχέση με τη συνολική δαπάνη προχωρεί σταθερά εύρυθμα. Όμως δεν θεωρούμε, λέτε στην έκθεση, ότι αυτό εξοικονομεί τα χρήματα του φορολογουμένου, ακριβώς όπως προσβεύουν τα θεσμικά οργάνα της Ένωσης. Πάρα πολύ κομψά λέτε. Όμως, τελικά δεν θα μπορούσατε να είστε πιο σπαθάτος όσον αφορά. Αυτή την πρακτική όσον αφορά την απεικόνηση της πραγματικότητας για τα συγκεκριμένα έργα. Θα ήθελα τη γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου, μια που εσείς είστε ε, κυρίως αρμόδιοι. Uh, ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Ναι, όντως δεν διακρίνει αυτή την περίπτωση μεγάλη διαφάνεια. Εκεί που έχουμε αυτού του είδους τις πιστώσεις, κάποιους ενδιαμέσους, είτε κρατικέ αρχέ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τελικά έχουμε αυτό το ραμασάζ το τέλο τη χρήσεως για να λιάνουμε αυτά τα κονδύλια. Αυτό είναι το καλό. Όμω, στην σύσταση υπερθυμών 3 λέμε ότι θα πρέπει να ε, έχουν περισσότερη διαφάνεια χρηματοδοτική μηχανισμοί από πλευρά των θεσμικών οργάνων για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Και βέβαια, μία από τις λύσεις θα ήταν να έχουμε διαφοροποιημένη δαπάνη για την πολιτική των κτηρίων να προκαθορίζονται τα ποσά που θα περάσουν μετά από τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Και όποτε έχουμε προκαταβολές για τα κτίρια, υπάρχει ο κίνδυνος στο τέλος της χρήσης, η προκαταβολή να μην αντικατοπτρίζει την πρόοδο του έργου. Εδώ όντως υπάρχουν ζητήματα. Ο πρόεδρος. σωστά, Αλλά εσείς υπερεκτιμάτε, υπερβάλλετε για κάποια κονδυλία. Μιλάμε για 30 ή 40 εκατομμύρια που καλύπτεται με το ραμασάζ. Εκπλήσουμε που δεν έχετε πιο κρυστάλλινη θέση ως ελληνικό συνέδριο. Θα μου δείτε κάποια έργα τα οποία θα πρέπει να τα έχετε εντάξει στον προπολογισμό. Και έτσι φύγεται το κύριο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Φύγεται πολύ το κύριο. Μια που είναι χρήματα τελικά των κρατών μελών εν μέρει. Άρα θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα προς μίμηση, να είναι υποδειγματική η κατάρτιση και η εκτέλεση του προπολογισμού. το εκλαμβάνετε ως ε, ψόγο αυτό που σας λέω. Με κάθε σεβασμό, κύριε Γκρέγκορ. Ναι, ναι, συμφωνώ, πρόεδρε. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να παρουσιάζουν τα ποσά στον προπολογισμό που σχετίζονται με την ε, πρόοδο, με την κατάσταση τέλος πάντων πρόοδο των εργασιών των κτηρίων. Και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό και λέμε ότι το χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση των συστάσεων ε, θέλουμε να καλύψει τα έργα που θα, που θα αρχίσουν μετά το τέλος του 19 και έτσι ελπίζουμε τα σχετικά προβλήματα να λυθούν. Ωραία. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να έχετε άλλη στάση ως ελεγκτικό συνέδριο. Κάνετε εκπτώσεις στη, στην αντίληψη τη ρεαλιστική των πραγμάτων. Γι' αυτό δεν είναι το καλύτερο για τα δημιουργικά Θέλει κάποιος το λόγο. Donc, je vais vous appeler dans l'ordre que j'ai cité il y a un instant, pour que vous puissiez nous dire comment vous percevez le rapport de la Cour. την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Κύριε εσείς σίγουρα δεν υπερβάλλατε στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Εκπροσωπείτε την ΙΝΛΟ, Τα έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μας ενημερώνετε αρκετά. Οπότε με την ιδιότητά σας ως ε, μέλος, ως βραχίων του προϋπολογισμού, κύριε Ελλήνους πώς βλέπετε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και το Ελληνικό Συνέδριο για αυτή την αξιόλογη ε, έκθεση. Πρώτα πρώτα Πρόεδρε να πω κάτι για το σχόλιο σας όσον αφορά την ενημέρωση προς εσάς, τη δική μας. Υπάρχουν κάποιες ε, δαπάνες για την ασφαλεία, τα συζητήσαμε το, το, το, το καλοκαίρι και ε, βεβαίω έχω κληθεί εδώ στην Επιτροπή όσον αφορά το γραφείο των ε, Παρισίων και τον Φεβρουάριο επίσης ευχαριστώ να έρθω και θα έχουμε το σημείο όπως το ζητήσατε από τη γενική μας ε, διεύθυνση. Τώρα, για να δούμε την, την έκθεση του συνεδρίου που μας προσφέρει ο κύριος Γκρέγκορ. Πρώτα πρώτα, από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης Ίνλο του Κοινοβουλίου, χαιρόμεθα να συμφωνήσουμε. Ορθώς θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διοργανική συνεργασία διαμέσου των ετών έχουμε βελτίωση τη επίδοσή μας σε αυτό. Ξεκίνησε η διαδρομή αρχέ δεκαετία του 90 για όλου του τόπου εργασία και δεν ήταν στο σημερινό, ε, στη σημερινή ποιότητα η συνεργασία οργάνωση, συναδελφικότητα, επίσημη και ανεπίσημη ταυτόχρονα από πλευράς τώρα του Κοινοβουλίου. Με χαρά μας παρατηρούμε ότι το ζήτημα της κυριότητος ή της ε, μισθώσεως των ακινήτων αναδεικνύεται στην έκθεση του συνεδρίου. 80% έχει κυριότητα των κτηρίων του το Κοινοβουλίο. Σε αποτέλεσμα των όσων αποφασίστηκαν από κλάση δημιουργική στα μέσα δεκαετία του 90. και επί μακρόν δεν είχαμε άλλη απόφαση για τη στρατηγική την ακολουθητέα. Επίσης, το 2010, τον Μάρτιο, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για πρώτη φορά ενέκρινε τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια. Στη συνέχεια αυτή η στρατηγική συγκεκριμενοποιήθηκε, διευκρινίστηκε με άλλες αποφάσεις του Προεδρείου. Μετά το 2010. Και φυσικά όλα αυτά υπευλήθησαν ένα αρμοδίο στην αρχή του προπολογισμού. Η στρατηγική προσαρμόστηκε, εξυγχρονίστηκε με απόφαση του Προεδρείου τον Απρίλιο του 2018 και ίσως θα θυμάστε την παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα τον Ιούλιο εδώ στην Επιτροπή σας όσον αφορά την ε, νέα τροποποιηθήσα στρατηγική η οποία σε μεγάλο βαθμό καλύπτει το στοιχεία που χρειάζονται που δεν εκαλύπτονται για τα κτίρια. Και ρυθμίστηκε διάφορα ζητήματα ευέλικτε δυνατότητε ε, συνάντηση για τιμέ διαλόγου προ το κοινοβούλιο. Θα έρθει πιο κοντά ε, στον κόσμο την ε, αναβάθμιση της ασφάλειας των κτηρίων και Α, κάτι που είπε ο κύριος Γκρέγκορ. Αλλά εδώ φύγει και η έκθεση τους νέους τρόπους, νέες μεθόδους εργασίας. Το Κοινοβούλιο εκπώνησε μία μελέτη το 2015. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, στο Άουρ και στο Μάρτενς ε, αυτή η μέθοδος θα έφερνε εξοικονόμηση 110 εκατομμυρίων ευρώ σε μία εικοσαετία με αυτές τις νέες μεθόδους εργασίας. Όμως, εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα το 2015. Πάντως τώρα η διοίκηση εφαρμόζει κάποια από τα στοιχεία εκείνης της ιδέας, εκείνης της πρότασης σε αυτά τα δύο κτίρια. Και υπάρχει ένας ε, ζωηρός διάλογος των ε, εμπλεκομένων ε, υπηρεσιών, με όσους ε, θα στεγαστούν σε αυτά τα κτίρια. Όσοι ήδη είναι εκεί, όσοι θα μετακομίσουν εκεί, καλύπτονται από αυτήν την συνεργασία. Ήδη έχουμε feedback ε, πολύ θετικό για το Martens. Πολύ πολύ θετικά τα μηνύματα όσον αφορά την εφαρμογή των νέων μεθόδων εργασία. Τώρα, κάποια άλλα στοιχεία που αφορούν ε, χρηματοδότηση, σχετικούς μηχανισμούς. Ο κύριος Κλέτη εδώ είναι ορμόδιος ε, γενικός διευθυντής, και και ε, Τώρα, για τους managers, για την υποβολή των εκθέσεων, συμφωνούμε. Πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Και πριν από μόλις να με χρόνο στο έργο για το ε, έχουμε εισαγάγει ε, κάποιο είδους μη γραφειοκρατική ε, ευέλικτη μορφή management. Θετικό κρίθηκε όλο αυτό. Ευχαριστώ μου δώσετε το λόγο πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Αυτός ο ε, χώρος συνεργασίας έχετε μπορέσει να υπολογίσετε την οικονομία χώρου και τις οικονομίες ε, χώρων γραφείου που έχουν επιτευχθεί. Απάντηση. Για να απαντήσω σε αυτή την ειδικευμένη σας ερώτηση, στην ε, στρατηγική κτίριων που ενέκρινε το Προεδρείο και που συζητήσατε κιόλας Ε, θελήσαμε να δώσουμε 10 με 12 τετραγωνικά μέτρα ανά εργαζόμενο, ανά πρόσωπο. Άρα κάθε γενικός διευθυντής, μάλλον κάθε γενική διεύθυνση, έχει την ικανότητα να καθορίσει με ποιον τρόπο θα εργάζεται. Ορισμένες γενικές διευθύνσεις θα κατευθυνθούν περισσότερο προς την κατεύθυνση ε, ατομικών γραφείων ή γραφείων που μοιράζονται δύο-τρία άτομα. άλλε ε, βάζουν σε κοινά γραφεία τέσσερις συναδέλφου, με μία ή δύο εξαιρέσει μετά όμως από αίτηση των ίδιων των υπηρεσιών λόγω ειδικών καθηκόντων όπως για παράδειγμα ανθρώπων που ασχολούνται με τις επικοινωνίες ή την ηλεκτρονική τεχνολογία Γενικώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί μεγάλους χώρους συνεργασίας όπου οι άνθρωποι δεν έχουν γραφείο διατεθειμένο ειδικά για αυτούς. Γραφείο με την έννοια του desk. Η γίνει προσπάθεια για το λεγόμενο νέο κόσμο εργασίας αλλά ε, οι απαντήσεις που λάβαμε από χίλιους περίπου εργαζομένους ε, στο κτίριο Μάρτινς ήταν πολύ θετική, διότι τους επέτρεψε καλύτερη χρήση των χώρων γραφείων που είναι διαθέσιμοι και επίσης ε, ενισχύθηκαν οι κοινωνικές πτυχές που ζήτησε το Προεδρείο. Δηλαδή κάποιες γωνιές όπου μπορεί κανείς να πιει ένα καφέ, μπορεί να ε, συναντηθεί ε, ανεπίσημα με άλλους και να συζητήσει και το καθεξής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κλετή. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι σε τρία θέματα. Την περιπλοκότητα της χρηματοδοτήσεως, την αναγκαία διαφάνεια και ειλικρίνεια και τέλος την αυ το αυξημένο κόστος των καθυστερημένων μισθώσεων. Πρώτα να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Γκρεγκόρ. Τα θεσμικά όργανα εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διαθέτουν αποδεσμευμένες πιστώσεις με τις οποίες να μπορεί κανείς να σχεδιάσει και να χρηματοδοτήσει για πολυετή περίοδο ανάγκες χρηματοδοτήσεως και cash flow για κάθε χρονιά. Αυτό δεν υπάρχει. Δεύτερο, όταν αρχίσαμε με το σχέδιο CAD δεν μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα. Επίσης, ως γνωρίζετε, σε κοινοβούλιο υπάρχουν προϋπολογισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται αναλόγως με τα έτη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Έχουμε προϋπολογισμούς, για παράδειγμα, για τα έτη των εκλογών που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, αλλά προσπαθούμε να παραμένουμε σε ένα πλαίσιο αυτό το οποίο προκαθορίζεται από τον τίτλο 5. Η περιπλοκότητα απορρέει από την χρήση αυτών των εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό, η περιπλοκότητα δεν κρίθηκε ως καλή ή κακή από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν θέλω να κάνω άλλους παραλληλισμούς, αλλά η χρηματοδότηση υπό δύσκολες ρυθμιστικές συνθήκες ένα έργο 430 εκατομμυρίων μέσα σε ένα προκαθορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτεί κάποιες καινοτόμες ιδέες. Και νομίζω ότι η περιπλοκότητα που ε, χρησιμοποίησαμε τελικά μπόρεσε να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε σωστά τα, τις δημοσιονομικές προκλήσεις κάθε φορά που ήταν δυνατόν να μην πληρώνουμε τόκους, αλλά πιο πολύ να κινητοποιήσουμε κάποια υπόλοιπα του προϋπολογισμού που δεν είχαν υπερτιμηθεί αρχικά. Το, το διευκρινίζω αυτό. Έχουμε κάνει έως τώρα 7 ραμασάζ, τα οποία μας επέτρεψαν να, ε, να εξοικονομήσουμε σχεδόν 98 εκατομμύρια ευρώ. Ε, πρόκειται για θέματα ειλικρίνειας, τα οποία απολύτως σεβόμαστε. Διαφάνεια και ειλικρίνεια όμως, ε, αυτή ε, γίνεται σεβαστή και με το ex post reporting στο, στην επίσημη εφημερίδα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δημοσιεύονται όλες οι μεταφορές. Κάθε φορά την μεταφορά του ραμασάζ με τη σχετική δημοσιότητα ε, δηλαδή δημόσιε συζητήσει, τις οποίες μετά ε, παρακολουθεί και εγκρίνει η Επιτροπή Προπολογισμών και μετά περιλαμβάνονται και ενσωματώνονται οι σχετικοί λογαριασμοί μέσα στο ε, έγγραφο. Άρα υπάρχει διαφάνεια και όταν εγκρίνεται και όταν τροποποιείται ο προπολογισμό. Και όταν εκτελείται. Υπάρχουν άλλωστε υποχρεωτικέ δημοσιεύσει μετά, και μετά την εκτέλεση των κονδυλίων. Αυτά σε ό,τι αφορά την διαφάνεια που κατά τη γνώμη μου γίνεται απόλυτα σεβαστή. Σε ό,τι αφορά την ειλικρίνεια υπενθυμίζω ότι οι γραμμές του προπολογισμού δεν υπερτιμώνται. Είμαστε ένα όργανο το οποίο ασκεί πολιτική δραστηριότητα η οποία κάποιες στιγμές μπορεί να οδηγήσει ώστε για παράδειγμα τα ταξίδια των ευρωβουλευτών να μην εξαντλήσουν τα προβλεπόμενα κονδύλια ή ε, τα επιδόματα για τους ε, συνεργάτες των βουλευτών να επίσης να μην εξαντληθούν. Αυτό το ραμασόδαν έρχεται σε 3%. 3 έως 5%. Δηλαδή πρόκειται για ένα ποσό σχετικά αμεληταίο διακόπτει ο Πρόεδρος. Επ' αυτού, κύριε Κλετή, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Αν δεν γίνει ραμασά στο τέλος του έτους, τι κάνετε. Εδώ επανέρχομαι στην ε, περιπλοκότητα που ε, ταυτόχρονα δίνει όμως και ένα στοιχείο ευκαμψίας, διότι ο δημοσιονομικό κανονισμός θα μας επέτρεπε να ε, δανειστούμε για την φάση της κατασκευής, άρα να πληρώσουμε τόκους σε όλη τη φάση της κατασκευής και βεβαίως στην φάση της επιστροφής του δανείου. Έχουμε λοιπόν μια δυνατότητα δανεισμού. Πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση πριν από την εκκίνηση του έργου, διότι δεν έχουμε ούτε πιστώσεις αιτήσει εγγεγραμμένες στον προπολογισμό, ούτε το ραμασάζ. Άρα η βάση της χρηματοδότησης είναι γραμμή του προπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από εμπορικές τράπεζες. Βεβαίως με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους. επιτόκιο 0,3% εάν χρειαστεί να δανειστούμε. Εκεί βρισκόμαστε. Εκτός αυτού υπάρχει ο μηχανισμός ε, που επιτρέπει να δίνονται κονδύλια για την κατασκευή, στη διάρκεια της κατασκευής. Δεν κάνουμε όμως προκαταβολές, δεν δίνουμε προκαταβολές, αλλά από τη στιγμή που έχουν πέσει τα μπετά, από τη στιγμή εκείνη οι πιστώσεις που δίνονται παραμένουν στην κυριότητα του Κοινοβουλίου. Αν έχουμε διαθέσιμα, διαθέσιμες πιστώσεις ή χάρη στο ραμασάζ έχουμε κάποια αποθεματικά, έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε στη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Στις εκθέσεις που συντάσσονται και στις ε, εκθέσεις που δημοσιεύονται στην, στο επίσημο έντυπο, όλα αυτά φαίνονται καθαρά. Δεν μπορέσαμε να πείσουμε το ελεγκτικό συνέδριο ωστόσο στο εξή για την αξιολόγηση ενός ενδεχομένου υπέρτερου κόστους λόγω των καθυστερήσεων και λόγω του γεγονότος ότι εξακολουθούμε να μισθώνουμε κτίρια, άρα πληρώνουμε μίστομα της τάξης των 14,3 εκατομμυρίων τον χρόνο και θεωρούμε εκεί ότι πρέπει να γίνει μια καθαρή διαφοροποίηση ανάμεσα στα, στο τελικό κόστος κατανάλωσης που είναι δάνεια ή αποσβέσεις αποτελέσμα χρήσεως δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να φαίνονται καθαρά οι τελικές δαπάνες είτε πρόκειται για μισθώματα είτε πρόκειται για ε, αποσβέσεις για την περίοδο που διανύουμε και που αποσβαίνεται την πρώτη μέρα της εφαρμογής. Και βεβαίως οι επενδύσεις αυτές παραμένουν στην κυριότητα των ε, Ευρωπαίων πολιτών. 430 εκατομμύρια, τα οποία έχουν εγκριθεί τώρα στην φάση της επενδύσεως πρόκειται για μια χρηματοδοτική ροή που προέρχεται από τον ε, Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δεν είναι όμως τελική δαπάνη με την έννοια ότι μεταφέρεται αμέσως στον ισολογισμό του θεσμικού οργάνου και επομένως στον ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φορολογούμενος πολίτης δηλαδή παραμένει κύριος υπό άλλη μορφή ούτως ή άλλως έχει καταβάλει τους φόρους του, παραμένει όμως κύριος του κτηρίου. Την ημέρα όπου θα αρχίσει να λειτουργεί το ΚΑΤ, δεν θα έχουμε πλέον να πληρώνουμε μίσθωμα και θα υπάρχει απόσβεση τη τάξη των 17 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο σε σύγκριση με το μίσθωμα, διότι η λουξεμβουργική κυβέρνηση υποστηρίζει το έργο και έχει ε, προσφέρει χαμηλότερα μισθώματα σε όλη τη φάση της σε όλη τη διάρκεια της φάσης της κατασκευής. Το ένα λοιπόν είναι μια τελική δαπάνη που είναι τα μισθώματα, το άλλο είναι δαπάνη επενδύσεως, όπου κύριος παραμένει αυτός που πληρώνει, δηλαδή ο φορολογούμενος πολίτης. Ευχαριστώ για τη ευκρινήσεις σας. η επιχορήγηση της λουξεμβουργικής κυβέρνησης ανέρχεται σε ποιο ποσοστό. Περίπου 50% του μισθώματος. Υπάρχουν ε, τρέχουν διάφορες μισθώσεις όπως το κτίριο Σούμαν το οποίο επιδοτείται περισσότερο ακόμη από τη λουξεμβουργική κυβέρνηση και το οποίο, γεγονός το οποίο επιτρέπει να παραμένει το μίσθωμα στα 14 εκατομμύρια αντί στα 22 που θα ενοχόταν. Κυρία Γουάρδια Ζαμπάλ, θέλετε να παρέμβετε. Ορίστε. Άκουσα την κύριε Λίνος. Αλλά ήθελα κάτι να πω το ότι αυτά που μας είπε δεν έχουν τόσο σχέση με την έκθεση, αλλά αυτά που είπε είναι θέματα κοινή αρμοδιότητα. Αξιόλογα τα σχόλια. θετικά κάποια που είπε και μερικά άλλα όμως όχι τόσο. όπως όλοι μας ε, ξέρει πολλά για πολλά πράγματα Οπότε για να δούμε αν χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο που μπορούμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, αλλιώς να έχουμε απλώς κάποιο διάβλο επικοινωνία, αλλά αν έχει κάτι να προτείνει θα μπορούσε να μα τα δώσει και εγγράφο το σωστό για το μέλλον το, το, κοινοβούλιο να μπορεί να προχωρήσει επί τη βάση όλων όσων γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ για την ευκαιρία να διευκρινίσω το θέμα αυτό. Όντω, Είχαμε πολλά αρνητικά σχόλια προτού α, μετακομίσουμε στο κτίριο Μάρτενσα. Υπήρξαν πολλέ ανησυχίε που εκφράστηκαν από την Επιτροπή Προσωπικού και από διάφορα συνδικάτα του προσωπικού. Νομίζω ότι και εγώ παρουσιάστηκα στην Επιτροπή Προσωπικού σε τρεις περιστάσεις προκειμένου να διευκολύνουμε μια ανοιχτή διεξαγωγή διαλόγου και να εξηγήσω και στην Επιτροπή Προσωπικού και στο προσωπικό που είχε ανησυχίες ότι συνολικά στη διαδικασία διαβούλευσης με τον κόσμο είχαμε διοργανώσει 190 συνεδριάσεις και συναντήσεις οι οποίες διοργανώθηκαν καταρχάς από την διοίκηση αλλά και από το προσωπικό των διαφορών μονάδων πριν μετακομίσουμε, μετά τη μετακόμιση που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του περσινού έτους. Άρα δεν έχουμε ακόμα κλείσει τα τέσσερα έτη μετά τη μετακόμιση, που είναι το σύνηθες χρονικό διάστημα μετά το οποίο κάνουμε μία αξιολόγηση. Και πάλι λοιπόν παρευρέθηκα μετά από πρόσκληση του, της Επιτροπής Προσωπικού ενώπιον της ε, Επιτροπής ε, και εκεί η Επιτροπή Προσωπικού διευκρίνησε ότι πλέον τα αρνητικά και επικριτικά σχόλια είχαν πάυσει. Φυσικά παρέμειναν κάποια ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την διαδικασία προσαρμογής η οποία την οποία περνάει κάθε κτίριο. Το κτίριο αυτό μιας και έχει έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα Υπάρχουν διάφορα στοιχεία σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό και άλλες τεχνικές περιγραφές, οι οποίες χρειάζεται να προσαρμοστούν. Ωστόσο, όλες οι κριτικές ε, για τους κοινού χώρους, για τα κοινά είχαν πλέον πάυσει. Όταν θα κλείσουμε με το καλό των τετραετία, θα κάνουμε πολύ πιο λεπτομερείς αναλύσεις των ε, ενδεχόμενων παρατηρήσεων. Αλλά και από δική μα πλευρά από την πλευρά τη ε, Γενική Διεύθυνση ΙΝΛΟ, χάρηκαμε ιδιαίτερα γιατί κάποιες ανησυχίε οι οποίες είχαν εκφραστεί εκ των προτέρων τελικά δεν ε, πραγματοποιήθηκαν, ήταν υπόστατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριο ε, Κρετή. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την αξιολόγηση που κάνετε σε ένα θεσμικό πλαίσιο πολύ περιπλοκό. Ίσως το λεκτικό συνέδριο όμως θα μπορούσε να κάνει συστάσεις για να αλλάξουμε το κανονιστικό πλαίσιο χωρίς να αγγίξουμε την ε, συνθήκη. Από ποια αρχή λοιπόν εξαρτάται ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε. Ε, δική σας ευθύνη ως ε, συνομοθέτη. Ένα από τα δύο θέματα είχαμε, ήταν η έλλειψη δυνατότητας ε, μίσθωσης. χωρίς σχετικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Το δεύτερο είναι τα σύμβερτα κεφάλαια. Και πάλι εδώ ο οικονομικός κανονισμός τα ορίζει αυτά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε μία κατηγορία πιστώσεων για τα πολυετή έργα σε ό,τι αφορά δεκαετία, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος, κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον κανονισμό και τελικά έχει ως αποτέλεσμα αυτό να προκύπτουν πολύπλοκες ε, υποχρεώσεις που ουσιαστικά στρεβλώνουν και τις θεμελιώδεις ε, αρχές του προπολογισμού, μα τότε θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός. Το ελεκτικό συνεδρίο και εσείς οι ίδιοι μας κάνετε συστάσεις για την τροποποίηση του κανονισμού και αν έχουν προβλεφθεί 40-50 ε, εκατομμύρια για παράδειγμα για το κτίριο κάτι στο Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, πρόβλημα, θεωρώ, να προσθεθούν στη φάση τη προγραμματισμού 42 εκατομμύρια τα οποία έτσι κι αλλιώ θα συσσωρεύονταν μετά. Και αυτό θεωρώ ότι ε, θα ήταν λογικό. Οπότε όταν λέτε ότι γλιτώνουμε τους τόκους, αυτό είναι καλό, αλλά φυσικά να σας πω ότι εφόσον είναι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που δανείζονται. Αυτοί οι τόκοι έχουν ε, και επιβαρύνουν τελικά και τον ευρωπαϊκό προβλαγισμό. Και να ακούσουμε τώρα λοιπόν, λέει ο πρόεδρο ε, τον κύριο Μουρίνιο και τον κύριο Μπέκε. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια. Και μια και έχει περάσει και η ώρα, αν θα μπορούσατε παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, από το Λουξεμβούργο. Να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το Ζαν 2, όπου επισημάνεται μια σημαντική καθυστέρηση από το Ελληνικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του έργου. Να πω ότι δεν συμφωνούμε με την αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική επίπτωση μια σκηνή από το Ελληνικό Συνέδριο, γιατί θεωρούμε ότι κάποια στοιχεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη, είναι κάποια στοιχεία ενδεχομένω ε, ε, έχουν ληφθεί υπόψη, αλλά χωρίς να υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού σε ό,τι αφορά την εγκατάλειψη, για παράδειγμα, του Ζαν λόγω του αμύαντου που υπήρχε εκεί. Και μας λένε λοιπόν, έχει ελευθερωθεί το έργο, θα μπορούσαμε να τα κινηθούμε χωρίς να χρειαστεί εγκρίστοση άλλου κτηρίου. Αυτό το έχουμε συζητήσει στο έπακρον μεταλλητικό συνέδριο. Αλλά η παράδοση του Ζαμονέ 2 με καθυστερημένο χρονικό ορίζοντα σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να αποπληρώνουμε και πιο αργά το μόνο 2. Άρα εδώ υπάρχει μια αντιστάθμιση, μια εξισορρόπηση. Είναι λίγο πιο περίπλοκτα πράγματα από ότι θα πίστευε κανεί ε, εκ πρώτη όψεω εξετάζοντα απλά τα έργα. Από την άλλη, χρησιμοποίησαμε και την καθυστέρηση αυτή για να βελτιστοποιήσουμε το έργο. Γιατί σε πρώτη φάση Είχαμε 3.040 ε, συναδέλφους αρχικά προβλεπόταν σαν γραφεία για 3.040 συναδέλφους, πλέον είναι 3.600 αυτοί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά επιμέρους στοιχεία, τα οποία ωστόσο διαμορφώνουν ε, με διαφορετικό τρόπο τον συνολικό πίνακα. Από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Αυτή η βελτιστοποίηση λοιπόν έγινε δυνατή και χάρη στην έγκριση των νέων τρόπων εργασίας σε ό,τι αφορά του μελλοντικού εργαζόμενου στο Ζαμονεδίο, προκειμένου να αποτελεί αυτό ε, ένα χώρο συνεργατικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπέ και ο κύριο Μουρινιό. Έχετε να σχολιάσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Νομίζω ότι σε ό,τι μα αφορά από πλευρά τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κτίριο στι Βρυξέλλε, πρόκειται για μια έκθεση η οποία είναι αρκετά ισόρροπη. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία αποτελούν βάσιμε κριτικέ και θα τα εξετάσουμε και θα τα επιλύσουμε και νομίζω τα δύο σχόλια τα οποία έχουν γίνει νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα λεπίσουμε με επαγγελματικό τρόπο να πω δύο λόγια μόνο για τους νέους τρόπους εργασίας. Άκουσα καλά τα σχόλια του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά προφανώ πρόκειται για μια έννοια η οποία είναι σε εξέλιξη. Μπορεί να χρησιμοποιούμε του ίδιου όρου και δεκαετίε, αλλά έχουν αλλάξει όλα αυτά και αλλάζουν στην ουσία του, στο εσωτερικό. Αυτό καταρχά. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι θα ήταν, δύσκολο, θα λάθος να το περιορίσουμε το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τι επιφάνειε εργασία. Εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε και να αποδείξουμε ότι είναι λιγότερα τα έξοδα και είναι λιγότερε η έκταση που χρησιμοποιείται. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο γιατί χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τρία στοιχεία τα οποία λειτουργούν καλά μαζί του. Κοιτάμε την απόδοση του προσωπικού, τα θέματα τη πληροφορική που θα επιτρέψουν σωστή συνεργασία και καλή και προφανώ και το κτίριο. Αυτά, Πρόεδρε. Αυτοί οι τρει όροι πιστεύετε ότι πληρούνται, λέει ο Πρόεδρο, ή είναι όροι οι οποίοι δεν υλοποιούνται στην ώρα του, ε, Κοιτάξτε, θα πρέπει να τεθούν όλα αυτά σε εφαρμογή και θα πρέπει να αλλάξουμε και τη συμπεριφορά του προσωπικού και των διαφορών γενικών διευθύνσεων σε ό,τι αφορά και τι διευθύνσει. Νομίζω ότι εκεί είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Η κυρία Λένοξ μα είπε ότι θα πρέπει να εισαχθούν όλε αυτέ οι νέε αυτές οι νέες μέθοδοι. Αλλά ουσιαστικά για να γίνει αυτό πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Όταν το έχουμε πετύχει αυτό, λοιπόν, όσο δεν το έχουμε πετύχει αυτό, Υπάρχει μία ε, εικονική μόνο αλλαγή, δεν είναι ουσιαστική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Φανούλης από το Συμβούλιο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω κι εγώ κάποια στοιχεία σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Μουλινιό. Όντως, δεν πρόκειται για μία άσκηση που έχει αποκλειστικά ως στόχο τη μείωση των τετραγωνικών μέτρων των γραφείων. Όχι, αυτό είναι πολύ πιο ευρύ ως project. Breaks, bytes, behavior. Αυτά είναι τα στοιχεία όπως τα αναφέρουμε ενδεικτικά. Να βρούμε δηλαδή μια συνολική λύση η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού και στο να μπορεί το προσωπικό να βρει τον χώρο που του χρειάζεται κάθε φορά για να εκπληρώσει τις ανάγκες τους. Είμαστε σε φάση πληθυντική. Δεν είναι ε, σε φάση ε, έγκαιρης ε, έγκριση. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται από όλε τι πλευρέ και θέλουμε να επισκεφτούμε το κτίριο αυτό για να διδαχτούμε προκειμένου να διαμορφώσουμε και εμεί τι καλύτερε λύσει εφαρμογή και να εφαρμοστεί αυτή η νέα αμα, έννοια με τις εμπειρίες των τελευταίων ετών. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα με τις συστάσει του ελεκτικού συνεδρίου ότι θέλουμε να αξιολογηθεί το έργο αυτό, αλλά θέλουμε και σε δύο χρόνια να πειραματιστούμε με διάφορους τύπους νέων, τόπων, νέων τρόπων εργασίας, ε, το Flex Desk για παράδειγμα, και άλλους ε, τρόπους ε, γραφείων, διαμόρφωσης γραφείων. Αυτά που ανέφερε η κυρία Λάινεξ. θέλαμε λοιπόν να τα κοιτάξουμε αυτά για να δούμε τελικά ποιο είναι το πιο κατάλληλο λύση. Και όλα αυτά σε ό,τι αφορά το activity-based working, εργασία βάση δραστηριότητα. Διαφορετικοί τύποι λοιπόν εργασία, όπου θα μπορούσαμε είτε να οργανώσουμε μία συνάντηση με όλα τα πληροφορικά εργαλεία τα οποία θα θέλαμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους τηλεδιάσκεψης, τηλεργασίες, τι θα σήμαινε αυτό και για τα bytes και η συμπεριφορά. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τελικά τη συμπεριφορά του προσωπικού, το οποίο πλέον δεν θα έχουμε υπό την άμεση εποπτεία μα. Πώ θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα τη εργασία σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είναι περίπλοκο το θέμα, προφανώ. Και να πω και δύο λόγια για το κτίριο Γιρόπα και τις συστάσεις ε, και τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν. Να μιλήσω στα αγγλικά, λέει η μιλητρία, μιας και οι σημειώσεις μου είναι στα αγγλικά. Όπω αναφέρεται λοιπόν στο έγγραφο, αλλά το είδα στην παρουσίασή σα, το κτίριο Europa παρέμενε εκτό του προπολογισμού του, εντό του προπολογισμού του, συγγνώμη, το οποίο προφανώ είναι προ όφελο του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Υπήρξε μια καθυστέρηση. Η καθυστέρηση όμω προέκυψε από απρόβλεπτου ε, παράγοντε. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Είχαμε καταρχά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η οποία άλλαξε με σημαντικό τρόπο το πεδίο εφαρμογή των κτηριακών έργων. Άρα, χρειάστηκε να εφαρμοστεί μία νέα μορφή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό προφανώς είχε θέμα, είχε αντικτύπο και στην Προεδρία και στο κτίριο. Ελευθεί υπόψη. Επίσης έγινε μια αγωγή στο πρωτοδικείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά έναν ε, από τους οτιτούντες ε, στον αρχικό διαγωνισμό. Και αυτό οδήγησε στην ε, καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση επίση τριών ετών σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, αλλά εκ παραλληλού δεν υπερβληθήκε ο προπολογισμό. Μείναμε εντό προπολογισμού, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα συνολικά. Επίση, Πολλά έχουμε να πούμε για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, κατά πόσον είναι περίπλοκοι ή απλοί. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απλοί και αυτό είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η τελική σύμβαση την οποία ψήφισε, συγγνώμη, υπέγραψε το Συμβούλιο με το κράτος του Βελγίου υπεγράφει το 2008 και φυσικά αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι το τι ίσχυε τότε, το 2008, από τον οικονομικό ε, κανονισμό θέμα, τότε οι διαφορετικές ε, οι πληρωμές αυτές ε, ήταν ε, δυνατές, υπήρχαν ως δυνατότητα, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα για τα δάνεια τότε, το 2008. Άρα χρειάστηκε να υλοποιήσουμε το έργο αυτό με τα μέσα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας τότε, το 2008. Και κάναμε ε, προκαταβολές, δώσαμε προκαταβολές, αλλά προς το βελγικό κράτος, όχι σε κάποιον σκοτεινό επενδυτή ο οποίος ε, πτώχευσε, όχι. Το βελγικό κράτος για μας ε, θεωρούσαμε ότι ήταν ένας έμπιστος εταίρος, εξακολουθεί να είναι έμπιστος εταίρος και γι' αυτό λοιπόν κάναμε την προκαταβολή σημαντικού ποσού. Αλλά Αυτές οι πρακταβολές είχαν ως αποτέλεσμα 10,3 ε, εκατομμύρια σε τόκους, το οποίο αφαιρέθηκε από το τελικό κόστος του κτηρίου και αυτό πάλι η προσφορά του Ευρωπαίου Φορολογούμενου θεωρούμε. Αυτά λοιπόν τα κάποια σχόλιά μου και τα κάποια στοιχεία που ήθελα να σας αναφέρω και να τα λάβουμε υπόψη. Πέραν αυτών όμως συμφωνούμε απόλυτα με τις συστάσεις του αλεκτικού συνεδρίου και θα συνεργαστούμε και με τα άλλα θεσμικά όργανα για να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Άρα λέτε ότι αυτό συμφέρει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Δεν ξέρω αν συμφέρει όμω τον ε, Βέλγο φορολογούμενο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πόσο περίπλοκη είναι η όλη διαδικασία με όλα αυτά τα διαφορετικά βήματα για να διευκολυνθούν οι καταστάσει αυτέ. αν ε, με καλούσαν σε συνέντευξη τύπου να εξηγήσω πώς ε, χρηματοδοτήθηκε το έργο, θεωρώ ότι θα δυσκολευόμουν. Αλλά, όπως λέτε, ακολουθείτε και τη νομική πραγματικότητα και τον κανονισμό. Από το ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριος Γιέννης έχει το λόγο. Ο κύριος Γιέννης, συγγνώμη. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριος Σπίας να μιλήσω για τα θεσμικά όργανα στο Λουξεμβούργο και το ελεκτικό συνέδριο όλος ιδιαίτερο όπως αναφέρεται στην έκθεση του κυρίου Γκρέκορ, τον οποίο και ευχαριστώ που υπογράμμισε τα καλά αποτελέσματα που πέτυχε το ελεκτικό συνέδριο τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους πετύχαμε τα καλά αυτά αποτελέσματα. Αλλά βασικό λόγο θεωρώ ότι είναι η καλή σχέση με το κράτο του Λουξεμβούργου. Και νομίζω ότι ακριβώ αυτή τη σύσταση θα δίναμε και στα άλλα θεσμικά όργανα να πετύχουν αυτή την άμεση και ειλικρινή σχέση με τα κράτη υποδοχή. Γιατί αυτό νομίζω ότι βελτιώνει και τι δυνατότητε που έχουμε στη ε, διάθεσή μα, αλλά και να σα πω και την διάθεση και την ε, καλές προθέσεις που υπάρχουν. Ένα δεύτερο σχόλιο τώρα που ήθελα να κάνω. μιας και αξιολογούμε τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τις πρακτικές αυτές, νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε αυτά σε καταναλογία. Στο ελεκτικό συνέδριο Δεν νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον αντικτύπο του Ραμασάζ. Κοιτάμε τι γίνεται σε βάθος χρόνου σε όλα τα έτη εφαρμογής του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μάλιστα, λέει Πρόεδρος, και ακούω πραγματικά έκκληση υπέρ του Ραμασάζ. Θα δυσκολευτείτε να μου αλλάξετε τη γνώμη. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλετε στο πρωτογενή προπολογισμό τα έξοδα αυτά και όχι να περιμένετε τώρα μασάζ για να εκτιμήσετε το κόστος. Αυτά ήθελα να πω εγώ και κατανοώ φυσικά την ε, ρεαλιστικό τρόπο που τα αντιμετωπίζετε αυτά. Αν τώρα υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο κανονισμού, θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες του κανονισμού για να ακολουθούνται οι σωστές και υγιείς ε, πρακτικές ε, του προπολογισμού. Ο κ. Κισελεύσκη από την Τράπεζα, την ΤΕΠ. Ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγγνώμη. Θα είμαι σύντομο, γιατί είναι θετικά τα αποτελέσματα, εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στα πλαίσια του ελέγχου αυτού σε ό,τι αφορά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έγιναν δεκτέ δύο συστάσει τη τράπεζα και που βελτίωσαν περαιτέρω τη διαχείριση. Ο νέο τρόπο εργασία αναφέρθηκε να σας πω ότι το 2018 και εμείς εισάγαμε ένα τέτοιο μηχανισμό, τον οποίο θα κληθούμε να αξιολογήσουμε το 2020, προκειμένου να καταλήξουμε στα σχετικά συμπεράσματα και να βγάλουμε πορίσματα. Επίσης, σημειώνουμε το ότι το Ελληνικό Συνέδριο σημείωσε με θετικό τρόπο την ε, προσωπικό και εξαντλητικό έλεγχο των ε, διαδικασιών για το κτίριο τη Φραγκφούρτη. Ευχαριστώ και λέει ο Πρόεδρο. Ε, ακούσαμε όλου του εκπροσώπου των διαφορετικών θεσμικών οργάνων. Να στραφώ τώρα προ του συναδέλφου. Μήπω έχουν αυτοί κάποια σχόλια να κάνουν, ούτε εσεί. Ο κύριο Γκριγκόρ, λοιπόν, για να ολοκληρώσει το θέμα. Uh, Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα σχόλια από τα διάφορα θεσμικά όργανα. Επιτρέψτε μου σύντομα λίγα τελικά σχόλια, αφού πρώτα συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ενέκρινε επισήμως την στρατηγική, το Προεδρείο του δηλαδή, και στην κατατιμωλία ε, διαδικασία συζητήσαμε αυτά για την λογιστική μεταχείριση της εκ των υστέρων διαφοροποίησης ε, το, για το κόστος των κτηρίων. Μακροπρόθεσμα είναι περίεργο ένας δημόσιος προϋπολογισμός να καλείται να χρηματοδοτεί τις ε, ε, επενδύσεις του μέσω διαμεσολαβητών. θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτούνται μέσα από τα πλαίσια του ίδιου του δημόσιου προϋπολογισμού. Αναφέρθηκα και στις συστάσεις που έχουμε περιλάβει στην έκθεσή μας του 2007, όπου είχαμε προτείνει να χρησιμοποιηθούν διαφοροποιημένες πιστώσεις ε, Τώρα για τα συγκεκριμένα έργα. Στις αρχικές μου παρατηρήσεις αναφέρθηκα σε απρόβλεπτες συνθήκες, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Συμβουλίου. Ανάφερα, ανέφερα και διάφορους λόγους καθυστερήσεων των επιμέρους έργων που ορισμένες φορές ξεφεύγουν από τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων εξαρτάται από τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη χώρα μέλος. Στην περίπτωση του Λουξεμβούργου ήταν θετική. Στην περίπτωση του Συμβουλίου η συνεργασία με το βελγικό κράτος δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Συνολικά θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό ότι μετά από την κατημολία διαδικασία με πέντε εκπροσώπους καταλήξαμε ότι θα βελτιωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης της κατασκευής των ε, κτίριων της Ένωσης και να υπάρχει και συγκρισιμότητα δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και ευχαριστώ πολύ και εσάς και τα ε, θεσμικά όργανα για τη σχόλιά τους. Φτάνουμε στο τέλος της ακουράσεως. Λέει ο Πρόεδρος, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση. Ευχαριστώ τον κύριο Γκρεγόρ και το ελεγκτικό συνέδριο για την ποιότητα του εγγράφου. Ευχαριστεί ο πρόεδρος και τους διερμηνείς που δέχθηκαν να παίξουν καθυστερήσεις για να μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε την ακρόαση για την κτηριακή πολιτική των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των διαφόρων θεσμών και συγχαρητήρια για τον άθλο που ε, επιτυγχάνουν να μπορέσουν δηλαδή να εργαστούν στη βάση νομοθετικών κειμένων που είναι περίπλοκα και όχι πάντοτε τόσο αυτονόητα. Για τι συστάσει που μπορούμε να κάνουμε, για να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό, μεταξύ άλλων, ώστε να διευκολυνθεί η εργασία των αρμοδίων, θα κατανοήσατε ότι πρωτίστως μας ενδιαφέρει ένας προϋπολογισμός που να αποδίδει με αξιοπιστία το τι πράττει η Ευρώπη είναι ο τρόπος μας για να συμβάλλουμε στην δημοκρατία και να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ευθύτητα στους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή να μην είναι κάποια πράγματα τα οποία ρυθμίζουν μεταξύ μα. Χαίρο για την προσπάθεια του Λουξεμβούργου, αλλά και για το Λουξεμβούργο έχει ενδιαφέρον που έχει τόσα πολλά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εγκατεστημένα στο υψίπεδο του Κίρσπερκ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ε, την ε, συμβολή σας. Αν κατάλαβα καλά το Λουξεμβούργο επιδοτεί ένα μέρος των μισθωμάτων, όπως και το ε, βασίλειο του Βελγίου, το οποίο υποκαθιστά εν μέρη ε, στα θεσμικά όργανα. Ε, η επόμενη συνάντησή μας θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου. Βεβαίω υπάρχει μια μικρή αβεβαιότητα σχετικά με την συνεδρίαση της 29η Πρώτου. Α, θα διεξαχθεί. Καλώ λοιπόν. 29 Ιανουαρίου μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου Προεκολογισμού. Σας ευχαριστώ που παραμείνατε έως τώρα και να συγχωρήσετε την Προεδρία που δεν επετάχυνε τις ε, ε, διαδικασίες αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας με όλους. Λίγη συνεδρίαση.